Ladies and gentlemen, dear colleagues, let us start. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Ένα. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τις εξής αλλαγές Πρώτον, το 7 θα το δούμε μετά το 23, μετά το 24, θα το δούμε μετά το 20 και μετά το 16 και το 26 αναβάλλονται. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχω καμία ανακοίνωση. Να πάμε στο σημείο 3. Σχέδιο σύστασης για την ενισχυμένη συνεργασία στους τομείς της δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εφαρμογής αποφάσεων σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας των διεθνών ζευγαριών ο λόγος στον εισηγητή. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι σε κάποια σύγχυση. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω πράγματα που έχουμε ξαναπεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τα υπενθυμίσω. Οι προτάσεις που θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση είναι μια καλή συμβαστική λύση για τις διαφορετικές θέσεις του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να αποφύγω πράγμα που έχω ξαναπεί να υποβληθούν τροπολογίες όσο και αν είναι καλή την πίστη ή θεμητές. Η διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε είναι διαδικασία διαβούλευσης. Αλλά αν αποστείλουμε τη θέση μας χωρίς πολλές αλλαγές θα είναι ένα τεκμηριωμένο ε, μήνυμα, μια τεκμηριωμένη θέση που θα αντικατοπτρίζει την ε, ακλόνητη θέση των ε, πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου για τις τροπολογίες. Να διευκρινίσω ότι οι διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις συνεχίζουν να εφαρμόζονται και να ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών, είτε συμβάλλονται είτε όχι, στην ενισχυμένη συνεργασία. Η διευκρίνηση αυτή είναι περιττή έτσι κι αλλιώς διότι αυτό είναι προφανές. Δεν υπάρχουν βεβολίες από καμία πλευρά, διότι είναι και συνέπεια της μη συμμετοχή ορισμένων κρατών στην ενισχυμένη συνεργασία. Κατά συνέπεια, εξυπακούεται. Άλλες τροπολογίες προβλέπουν ένα ορισμό για κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην ε, διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά το κείμενο για το εφαρμοστέο δίκαιο για τα διαζύγια και την ε, διέρεση των περιουσιακών στοιχείων του 2010 ούτω ή άλλω καθορίζει τα συμμετέχοντα κρατημέλη, οπότε και πάλι δεν υπάρχουν ε, αμφιβολίε ή απορίε. Έτσι κι αλλιώ οι κανόνε δεν ισχύουν για τα κράτη που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, στη δικασία αυτή. Η αναγνώριση των διοικητικών εγγράφων πρέπει να γίνεται με τον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και θα είναι απαραίτητη εφόσον δεν υπάρξει εναρμόνιση των εθνικών οικογενειακών δικαίων, κάτι που τόσο άλλως δεν είναι ο στόχος των διαφορετικών προτάσεων. Έτσι ούτως ή άλλως τα κράτη-μέλη που δεν ε, αναγνωρίζουν το σύμφωνο συμβίωσης και δεν μπορούν να εκδικάσουν ε, κάποια διαφορά που μπορεί να προκύψει στο έδαφο του, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναθέσουν ε, ή μπορούν να αναθέσουν την υπόθεση σε μια δικαιοδοσία άλλου κρατουμένου που αναγνωρίζει τι συμβάσει αυτέ. Είναι σαφέ. Όπω το είχα λοιπόν προτείνει όταν είχαμε την πρώτη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων συνάδελφοι, είμαι πρόθυμο να δεχτώ αλλαγή στο κείμενο που μιλά για την αιτιολόγηση, την ε, ακριβή αιτιολόγηση που θα συμπεριληφθεί ε, στην τελική έκθεση μετά την ψηφοφορία μας, ώστε να μην γίνεται μνήα των κρατών που ε, προέβαλαν το δικαίωμα άρνηση κυρίας, προκειμένου να παραμένουν δηλαδή ανώνυμα. Θα έλεγα όμως να μην το λάβουμε υπόψη, συνάδελφοι, παρόλο που σέβομαι πολύ τις απόψεις σας, να μην λάβουμε υπόψη τις τροπολογίες αυτές, διότι είναι τροπολογίες, πώς να το πω, καλοπιστικές. και μπορεί να καθυστερήσουν την έγκριση της έκθεσης. Και να στερηθούμε για πολύ καιρό ένα κείμενο που ε, διαπραγματεύτηκαν τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Είναι κάτι που μπορεί να βλάψει τους Ευρωπαίους πολίτες εφόσον καθυστερήσουμε Και βεβαίω τι οικογενειακέ καταστάσει και τι περιπτώσει ανθρώπων που δεν έχουν κάποια εύκολη, εύκολο τρόπο να εκδικαστεί η υπόθεσή του. Διαφορετικού πολίτε από διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω το εξή. Να διευκρινίσω ότι για το σημείο 3 για την ενισχυμένη συνεργασία το Κοινοβούλιο δίνει τη συνένεσή του Δηλαδή να ανατρέξει κανείς την ενισχυμένη συνεργασία. Στην ουσία της εκθεσής μου δηλαδή. Ξέχασα να το αναφέρω, με συγχωρείτε και ακόμα μια φορά θερμές ευχαριστίες. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν παρατηρήσεις, δηλώσεις. Κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη που ήρθα στο τέλος της παρέμβασης του εισηγητού. Θα ήθελα εκ μέρους της ε, Ευελίνα Γκέπχαρτ που είναι ισχυώδης εισηγητρία να σας ε, αναφέρω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Δυστυχώς προσγειώθηκε αργά οπότε δεν θα μπορέσει να είναι στην αρχή της συζήτησης μαζί μας και γι' αυτό ζητώ και εκ μέρους της συγγνώμη και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ για να διαβάσω την δική τη παρέμβαση. Δεν την προτίμασα εγώ δηλαδή. Η κυρία Γκέπχαρτ χαιρετίζει την νέα πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για, ε, ε, για τι σχέσει συζύγων. Μιλάμε για 18 κρατημέλη τα οποία μπορούν να υποφεληθούν από την ε, ε, καλύτερη συνεργασία για, την, ε, για το συγκεκριμένο νομικό πεδίο. Μιλούμε για σαφείς κανόνες και προτάσεις που θα δείξουν στους πολίτες μας ποια είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για αυτούς. Μιλούμε για τα κυβερνήσει τώρα των 11 κρατών μελών που μέχρι τώρα δεν έχουν συμφωνήσει για την ενισχυμένη συνεργασία και τους ζητούμε σύντομα να συμβάλλουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τον τομέα αυτό. Επίσης, ως προς αυτό υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα. Επειδή αυτά τα 16 εκατομμύρια διεθνών ζευγαριών δεν πρέπει να τα αφήσουμε με ασάφεια σε ό,τι αφορά το πιο εφαρμοστό δίκαιο μπορεί να βγει τη δική τους περίπτωση. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ε, απέχουμε από την ψηφοφορία για το κείμενο αυτό και σε ό,τι αφορά τις σχέσει, ε, ε, σχέσεις ε, θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη που δεν τι γνωρίζουν να πάνε στο άρθρο 9, παραγράφος 1 για τις του συγκεκριμένου κανονισμού για τις κατεχωρισμένε σχέσεις. Η σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2011 ουσιαστικά ενισχύεται και πάει ένα βήμα παραπέρα με, τη νέα αυτή πρόταση. Γίνεται εποχή συγκεκριμένη, γίνονται Υπάρχουν και οι νέες τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την, ε, το εφαρμοστέο δίκαιο. Και, και αυτό θεωρεί η κυρία Γκέφχαρτ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό νέο, νέο στοιχείο. Υπάρχουν νέες δομές στις ε, νέες αυτές προτάσεις που ε, ουσιαστικά δεν ε, που ουσιαστικά αντιμετωπίζει την ε, διακριτική μεταχείριση απέναντι στις καταχωρισμένες ε, σχέσεις. Υπάρχει δηλαδή εξίσωση. Δεν φροντίσαμε να, δεν έχουμε, να υποβάλουμε τροπολογίες ως προς την πρόταση αυτή. Αυτά πρόεδρε και ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε. Ο κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν καταστάσεις ε, ανθρώπινες που θα πρέπει να διευθετηθούν όπως οι διάφορες ενώσεις και η νομική τους κατάσταση. Αλλά κύριε Καβαντά, δεν συμφωνώ ότι πρέπει να απαλληφθούν οι τροπολογίες. Βρίσκω ότι θα έπρεπε να υπάρξουν τροπολογίες για να καθοσυχαστούν κάποια κράτη. Πολύ λίγα είναι τα κράτη που θέλουν έτσι και να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, οπότε ακριβώ αυτέ οι τροπολογίε μπορούν να καθησυχάσουν και να διασκεδάσουν τι ανησυχίε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν δούμε το σχέδιο έκθεση για την κατάσταση του γάμου και το καθεστώ του γάμου, η τροπολογία 8 περιλαμβάνει την εξή φράση. Αμοιβαία αναγνώριση των διοικητικών εγγράφων που δεν μπορεί να αντιφάσκει με την αρχή τη επικουρικότητα. Αυτή είναι μια υπενθύμηση που θα μπορούσε απλώς να καθησυχάσει. Βέβαια, το να λέτε ότι δεν χρησιμεύει σε τίποτα, το βρίσκω λίγο εύκολο να υποθεί. Είναι κρίμα μια μνήμα που μπορεί να καθησυχάσει τα κράτη να μην περιλαμβάνεται. Ο ισχυρό κανονισμό δεν μπορεί να επιβάλλει στα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν το εθνικό του δίκαιο, το εθνικό οικογενειακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτο που διέπει το γάμο. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να καθησυχάσει κάποια κράτη. Υπάρχει μια ανάλογη τροπολογία για τα άλλα κείμενα, για τι κατακεγραμμένε, τι καταχωρισμένε ενώσει. Βρίσκω κρίμα να πετάξουμε αυτέ τι τροπολογίε οι οποίε θα ικανοποιήσουν τι προσδοκίε πολλών κρατών και ολοκληρωμένων πολιτών. Δηλαδή, θέλουμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διάθεση να παρέμβει στο οικογενειακό δίκαιο, αλλά προσπαθεί να ε, επιλύσει συγκεκριμένε περιπτώσει συγκεκριμένων ανθρώπων. Ευχαριστούμε, κύριο Βίλαντ. Ευχαριστώ. Η πρόταση του συναδελφού Τζαμπάτσκι για την αναβολή των συζητήσεων. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, δεν είπε ο συνάδελφο Καβάντα τίποτα και ο συνάδελφο φω και αυτό δεν μπορούσε να έρθει από την αρχή και μου ζήτησε να πω κι εγώ κάποια πράγματα εκ μέρου του. Η ψηφοφορία για την ενισχυμένη συνεργασία σε κάποια κράτη-μέλη για τις ε, περιουσιακές σχέσεις ε, των ε, γάμων και των καταχωρισμένων σχέσεων θα πρέπει να γίνει αύριο. Το κείμενο για τις καταχωρισμένες σχέσεις έχει μια ρήτρα στο άρθρο 9 παράγραφος 3 όπου προβλέπεται ότι τα δικαστήρια ενός κράτους μέλους που δεν γνωρίζει το θεσμό αυτό, αυτής της καταχωρισμένης σχέσης μπορεί να αρνηθεί την εκδίκαση της υπόθεσης. υπάρχουν και οι εθνικές ε, αναγνώριση σχετικά και δεν νομίζω ότι αυτό που αναφέρεται στο κείμενο είναι σκόπιμο να ισχύσει. Υπάρχει μια γνωμοδότηση από την ε, Υπηρεσία Δημιουργικών Δικαιωμάτων που λέει ότι και οι δύο προτάσεις λόγω της διακριτικής μεταχείρισης δεν θα πρέπει να ε, διαχωριστούν. Γιατί το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και γι' αυτό θα θέλαμε να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα και είναι καλό σκόπιμο να ψηφίσουμε άμεσα έτσι ώστε ο φάκελος αυτός να μπορέσει να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της Ολλανδική Προεδρία. Επίσης να τονίσω ότι λόγω ακριβώς της ειδική νομικής βάσης της παραγράφου 81.1.3 δεν βρισκόμαστε σε, σε, σε τομέα ε, συναπόφασης και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ε, στο κείμενο του ε, Συμβουλίου. Υπάρχουν λίγες τροπολογίες και αυτό δείχνει ότι το κείμενο αντικατοπτρίζει τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο συνάδελφος Φως ε, συμφωνεί με τις τροπολογίες Κομοντίνη, Σάιρς και Σφιεύκα και δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει, ε, να υπάρξει περαιτέρω αλλαγή του κειμένου και η προτεραιότητά μα θα πρέπει να είναι γρήγορα να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και να ολοκληρωθεί το πακέτο αυτό. Αυτά και ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει να σχολιάσει ο εισηγητής. Όχι. Απλώς ε, καταγράφω όλα τα σχόλια πολύ ενδιαφέροντα αυτά που άκουσα. Αλλά θα ήθελα να επανεπισημάνω αυτά που ανέφερα προηγουμένως και να σας ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα ψηφίσουμε για το σημείο αυτό, παρά το γεγονός ε, ότι έλαβα ενημέρωση ότι ο κύριος Τζαμπάσκι ήθελε να προτείνει να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Δεν είναι όμως εδώ. Ίσως αύριο το πρωί να επανέλθουμε σε αυτό. Σας το λέω για να μην σας έρθει απότομα. Σε αυτή τη φάση πάντως, για την ώρα, ψηφίζουμε κανονικά αύριο κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασής μας το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ. Βάσει της τροποποιημένης ημερήσιας διάταξης, τώρα θα πάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης ε, που... που αφορά τη μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμοδιότητες έως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων της. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω ότι είμαστε ήδη στο δεύτερο στάδιο της ε, μεταρρύθμισης ε, του ε, Δικαστηρίου της Ένωσης. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να καταργήσουμε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης σε συνέχιση της απόφασης που λάβαμε πέρσι. Υπάρχει τριμερής διάλογος κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, υπήρξε κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας στο Στρασβούργο και υπήρχαν δύο ζητήματα τα οποία χρειάστηκε να συζητήσουμε το πρώτο αφορούσε την νομική βάση και το δεύτερο την ε, διατήρηση ή μη ε, ενός άρθρου που αφορούσε τα εξειδικευμένα δικαστήρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδους συζητητής που ήταν εκεί ε, ήταν και πολύ μάλιστα, ε, για τη νομική βάση ήθελε το Συμβούλιο να μην αναφέρεται το άρθρο 256α. Τελικά συμφωνήσαμε να το διατηρήσουμε γιατί το 256 δεν είναι νομική βάση, αλλά οριοθετεί κάπως ε, την ε, δουλειά των συνομοθετών. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μην το καταργήσουμε και επειδή είχαμε εμεί ψηφίσει ήδη ούτως ή άλλως ε, τη διατήρηση του άρθρου αυτού, 256.1, αποφασίσαμε να το διατηρήσουμε. Επίσης ψηφίσαμε υπέρ την κατάργηση της δημιουργίας της δημιουργίας ε, ε, εξειδικευμένων δικαστηρίων ε, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην χρειάζεται, αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να χρειαστεί. Σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον να υπάρχει ήδη αυτό το άρθρο στον κανονισμό. Εν τη σοφία του λοιπόν το Κοινοβούλιο αποφάσισε να διατηρηθεί αυτό το άρθρο αν μία μέρα υπάρξει ανάγκη να ε, συγκληθεί ένα εξειδικευμένο δικαστήριο. Συμφωνήσαμε και σε αυτό με το Συμβούλιο. Ε, το ε, δικαστήριο ήταν επίσης παρόν, εκπροσωπείτο, οπότε ήταν τετραμερής, όχι τριμερής διάλογος. Αύριο θα ψηφίσουμε και αν ε, ε, όλα πάνε καλά μπορούμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί οι εννέα δικαστές που βρίσκονται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης θα ε, μεταβούν στο Γενικό Δικαστήριο και την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό. Οπότε καλό θα ήταν να αναλάβουμε αυτή την επίσημη απόφαση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές θα προτιμούσαμε τον Ιούνιο για να δοθεί η δυνατότητα ε, στα όργανα της Ένωσης να οργανωθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα απλώς να επανεπισημάνω τη δική μου θέση για την παράνομη κατάργηση ε, του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, γιατί δεν έγινε αξιολόγηση αντικτύπου, δεν έγινε ανάλυση του κόστος, καμία διαβούλευση με τους ε, δημόσιους υπαλλήλους και τους ε, δικαστές, ενώ έχουμε νέα, νέους, νέα είδη διακυβέρνησης και νέους τρόπους διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ποια θα ήταν η άποψή σας εσάς, αν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποφάσιζε, χωρίς τη γνώμη σας, την κατάργηση της γραμματείας, για παράδειγμα. Θα ήθελα, παρακαλώ, πριν κοιμηθείτε το βράδυ, να το σκεφτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, άλλες παρατηρήσεις? Δεν το νομίζω. Θα ψηφίσουμε για αυτό το σημείο αύριο. Συνεχίζουμε. Unfortunately for item number... Δυστυχώς, δεν είναι εδώ η κυρία Χάουτελα που είναι η για το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Μήπως γνωρίζει κανείς ε, από εσά ε, πού είναι. Όχι, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. can, uh, I am deal with this item. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στην νομική υπηρεσία για το θέμα αυτό. Ο κύριος Γκουίντο Ρίτσι είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια αναδιατύπωση και αφορά την προστασία από τις συνέπειες εξοεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μία τρίτη χώρα. Η αναδιατύπωση, η πρόταση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της προσαρμογής κάποιων διατάξεων πολύ τεχνικών αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, ε, υπήρξε μία περίπτωση όπου η ομάδα διαβούλευσης ε, της νομικής υπηρεσίας δεν μπόρεσε να δώσει ε, τη γνωμοδότησή της για την αναδιατύπωση αυτή. Ξέρετε ότι πρόκειται για μία συμφωνία αυτοπεριορισμού κάποιων προνομίων των συνομοθετών για να μπορέσουν να είναι πιο ευανάγνωστες ε, ε, κάποια, κάποιες νομοθετικές πράξεις. Αυτή η συμφωνία προβλέπει ότι μία γνωμοδότηση των τριών νομικών υπηρεσιών Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου ε, πρέπει να γίνει πριν από την νομοθετική πράξη ώστε να εξασφαλιστεί στο συνομοθέτη ότι το εγχείρημα της αναδιατύπωσης τεχνικώς ήταν σωστό και ότι δεν υπήρξε τεράστια και ουσιαστική αλλαγή στην ίδια την νομοθεσία. Αυτή τη φορά όμως οι νομικές υπηρεσίες δεν συμφώνησαν ε, γιατί το Συμβούλιο διαφώνησε όσον αφορά τη νομική βάση, ε, σας το έχω ξαναεπισημάνει ε, αυτό. Η, τα, υπόλοιπα όργανα όμως... Ε, πίστευαν ότι δεν ήταν τεχνικό το θέμα, δεν ήταν απλή κωδικοποίηση, αλλά ήταν θέμα ε, για, τον, ε, για τους συνομοθέτες. Οπότε υπήρξε και μία ομάδα ε, συμβουλευτική ε, η άποψή μας είναι κατόπιν ε, των εργασιών μας ότι δεν μπορούμε να ε, τοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να θεωρηθεί όχι αναδιατύπωση το συγκεκριμένο θέμα αλλά να ακολουθηθεί τακτική συνήθις διαδικασία που ακολουθείται για τέτοιου είδους προτάσεις. Ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις αν έχετε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρούτσι, από τη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μήπως θέλετε να πάρετε το λόγο? Doesn't seem to be the case. Μάλλον όχι. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις? Okay. We have thereby finished with uh, point number Τελειώσαμε λοιπόν με το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης ε, και πρέπει να διακόψουμε λιγάκι μέχρι τις 5 για να συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών στις 5 γιατί έχουμε κάποιους προσκεκλημένους για τις περιπτώσεις ε, ασυλίας. Οπότε διακόπτουμε μέχρι τις 5. Ευχαριστώ.